Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Υπέροχη χειρονομία και ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρίαση με αυτή την πανέμορφη εικόνα. Αν δεν έχετε αντιρρήσει προς την ημερήσια διάταξη, ας την εγκρίνουμε με μία αλλαγή που έγινε κατέ της πολιτικής ομάδας και που ζήτησε να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Vous avez été averti ce Άλλωστε ενημερωθήκατε γέρος από το πρωί. Παρακαλώ λοιπόν οι καθυστερημένοι να σπεύσουν να εγκατασταθούν. Έγκριση ημερήσια διάταξη το τελειώσαμε. Ανακοινώσει του Προέδρου θα τι βρείτε στο κομπούνιου. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης ε, της 8ης Μαρτίου. Ως ήθιστε, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα τα πρακτικά κατά το πέρα συνεδρίαση εφόσον δεν έχουν υποβληθεί παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οπότε περνάμε αμέσως στο σημείο 10. Την ώρα της ψηφοφορίας κατέφτασε και η Μπάρμπαρα, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε με την έκθεση της Αν Γένσεν, η οποία απουσιάζει. Non, elle ne vient pas, donc on peut... Θα έρθει? Όχι, ούτε καν. Οπότε ξεκινάμε. Sur le rapport de Anne Jensen. Πάτε την κάρτα ψηφοφορία σας, <clears throat> πάτε τον την κάρτα σας, εκτός από τον κύριο Ρικέ φαντάζομαι, για την έκθεση αυτή της κυρίας Γέμσα. λοιπόν, τώρα διανέμονται οι κατάλογοι ψηφοφορίας. Περιμένουμε δύο λεπτά για να διανεμηθούν οι κατάλογοι ψηφοφορίας. Εντάξει. Όλοι έχετε τον κατάλογο ψηφοφορία σας. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Τροπολογία 3, Αντρέασεν. Η εισηγήτρια κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές απέριπτε. Τροπολογία 9 της Γκουε, Η συγγήτρια κατά. Ψήφι υπέρ. Κανείς. Κατά. Όλοι. Από χε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 Παξάς. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. 10, 11, 12, 13, 14 όλες μαζί. Μπορούμε. Όχι. Μάρτα. Εγώ θέλω την τροπολογία Πάξα να ψηφιστεί χωριστά. Ευχαριστώ. Τροπολογία 10 Παξά. Ψηφίπε. Κατά. Μα πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογίες 11, 12, 13 και 14, πόρτας και κλούτ. Όλες μαζί ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία δια της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Από τρεις ψήφι κατά, τρεις ημίς. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15, Αντρέασεν. Κατά εισηγήτρια. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. αποχέ, Απορρίπτεται. 16 Παξά. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Α, μία ψηφο, Κατά. Αποχέ. Δεκτή. Αιτιολογικέ σκέψει. 4. Ε, η συγγήτρια κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία είναι τη εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλύπτει λοιπόν την τροπολογία 5. 6. Ανδρέασεν. Η σύντρια κατά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αν μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί την 7 και 8, πόρτας και κλούτ, κατά η σύντρια, ψηφί υπέρ. Κανείς, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία. κατά. Ο Τζέμς είναι κατά. Ναι. Δικαίωμά σας. Αποχές. Μία αποχή. Εντάξει, άλλη ενέκρινα Ωραία. Τι άλλο έχουμε να ψηφίσουμε. διορθωτικός προϋπολογισμός υπαριθμών 1 της Φραντσέσκα, χωρίς τροπολογίες. Έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Τέσσερις πλήφη κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγγέκριτε, Συγχαρητήρια. Φραντσέσκα. Για το σημείο 11 δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα μεταφορά πιστώσεων. Σημείο 12. Ο Ζουζέ Μανουέλ έχει εδώ ένα ένα, μια μεταφορά πιστώσεων και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η... πρόκειται για τροποποίηση δύο θέσεων ΑΕΣΤΕ σε θέσεις ΑΝΤΕ. Πρόκειται για δύο περίπου εκατομμύρια, αλλά έχουμε κάνει διάφορες αλλαγές στο οργανόγραμμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Στις 28 τροπολογίες έχουν εγκριθεί για, αυτά τα, για αυτές τις αλλαγές και αναρωτιέμαι αν αυτή η αλλαγή των θέσεων ΑΕΣΤΕ σε θέσεις ΑΝΤΕ μήπως θα μπορούσε να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2013 και κατά πόσο είναι κατεπίγουσα αυτή η πρόταση. Θα ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα προτού δώσω την θέση μου για την ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή άραγε για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Λαμασούρ εκπροσωπεί κάποιο στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, παρακαλώ. Μπορείτε να παρουσιαστείτε. Γιώχανης Κέντ. Είμαι επικεφαλής μονάδος υπολογισμού στην ΟΚΕ. Και η πρόταση τροποποίησης του οργανόγραμματος είναι κάτι που θα προτιμούσαμε να λάβει χώρα μέσα στο 2012 αντί να πρέπει να περιμένουμε ως το 2013. Και όπως αναφέρεται στο οικείο έγγραφο, πρόκειται για διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες. Θα προτιμούσαμε να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ήδη μέσα στο 2012. Αυτό μπορώ να σας πω. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος Λαμασού. Κύριε κύριοι, Πρέπει να έχουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι και μια μικρή τροποποίηση ούτως ή άλλως, οπότε εγώ προτείνω να υπάρξει θετική ψήφος για τη μετατροπή δύο θέσεων ΑΕΣΤΕ σε θέσεις ΑΝΤΕ. Ευχαριστώ, Λεωπρόεδρος υπέρ αυτής της μεταφοράς που υποστηρίζει ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Κατά. Παρά. Ναι. Τρεις ψήφοι κατά. Αποχές. Ωραία. Έχει εγκριθεί. Δεν έχουμε άλλες μεταφορές πιστώσεων για τον κύριο Φερνάντες. Και δεν έχουμε κάποιο φάκελο σήμερα για την πολιτική κτηρίων. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τέρμα οι ψηφοφορίες λοιπόν. Κυρία Χολμάιερ, χωρίς να της έχει δοθεί ο λόγος, εκτός μικροφώνου. Μια παρατήρηση μονάχα για τις ε, προβλέψεις του, της κτηριακής πολιτικής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα που ίσως, που ίσως θα ήταν πιο πρόσφορο να μετατρέψουμε τις παρεμβάσεις αυτές σε λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στην αρχή πάλι, στο σημείο 4 και δίνω το λόγο στην Αντιπρόεδρο Γιούτα Χάουγκ. Αφήνω την Πρόεδρε, μάλλον στην Αντιπρόεδρο Γιούτα Χάουγκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε λοιπόν στο σημείο αυτό. Ο πρόεδρος μας πάει να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Εμείς φανταζόμαστε ότι το κάνει για να υποστηρίξει τον τωρινό πρόεδρο της Γαλλίας. Σημείο 4. Έχουμε την έκθεση Giovanni Lavia για τον τρίλογο που αφορά τον προπολογισμό 2013. θα ξεκινήσει και ξεκίνησε ήδη μάλλον στην αρχή αυτή τη εβδομάδα. Τζοβάνι, έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 26 Μαρτίου, δηλαδή στις αρχές της ε, τρέχουσας εβδομάδας, έγινε ο ερηνός τριμερής διάλογος. Στην ουσία Πρόκειται για μια συνάντηση ανάμεσα στην Δανική Προεδρία και το Κοινοβούλιο, την παρουσία φυσικά της Κομισιόν. Η Δανική Προεδρία μέσω του Υπουργού Νικολάη Βάμεν, που είναι ο Υπουργό για τι ευρωπαϊκές Υποθέσει, υπογράμμισε Ποια είναι τα κεντρικά σημεία που προκύπτουν από τα πορίσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές του προπολογισμού για το 2013 που υιοθετήθηκαν από το ΕΚΟΦΗΝ στις 21 Φεβρουαρίου. Στην ουσία το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη για έναν ρεαλιστικό ε, προϋπολογισμό έτσι ώστε οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές να αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες που θα πρέπει που σημαίνει δηλαδή έλεγχο των δαπανών. Επιπλέον το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να προσέξουμε πολύ το επίπεδο των ραλ. Επιπλέον το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες πληροφορίες για το επίπεδο των πληρωμών και για τις προβλέψεις ε, εκτέλεσης του προϋπολογισμού για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και επιπλέον ε, τόνισε και μάλλον εντόπισε και αυτό το υποβάλλω ε, στην προσοχή της Προέδρου της Επιτροπής μας ότι θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη η χρηματοδότηση των ε, διαφόρων οργανισμών. Εξάλλου υπογράμμισε ότι χρειάζεται μία συμφωνία για την επιπλέον χρηματοδότηση με 360 εκατομμύρια του προγράμματος ITER. Εγώ στο όνομα του Κοινοβουλίου τόνισα ποια ήταν τα κύρια στοιχεία που προέκυψαν από τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια του Στρασβούργου και άρα στο τέλος καταλήξαμε συμφωνώντας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Όπως προτάθηκε και στον τριμερή διάλογο θα γίνουν άλλοι δύο στις 9 Ιουλίου και στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τη θέση του για το προϋπολογισμό την 30η ε, εβδομάδα. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η συνδιαλλαγή θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στις 24 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη μέρα μετά από την ψηφοφορία που θα κάνουμε για τη θέση του Κοινοβουλίου και τη 13η Νοεμβρίου. Όσον αφορά την ε, συνδιαλλαγή, θα έχουμε 26 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 9 Νοεμβρίου ελπίζουμε όχι όλη τη νύχτα της 9ης προς την 10η Νοεμβρίου την, στο Συμβούλιο με δύο τριμερείς διαλόγους 31 ε, Δεκεμβρίου και 7 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο συμφωνήσαμε και θα σας ενημερώνουμε στη διάρκεια της διαδικασίας. Δεν έγιναν πιο λεπτομερείς ε, επαφές ως ήθιστε σε αυτό το πρώτο τριμερή διάλογο. Ευχαριστούμε Τζοβάνι. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα είναι όχι ακριβώς τρίλογος, αλλά μονόλογος. Δηλαδή κάθε πλευρά θα παρουσιάσει τη θέση της, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία μεταξύ μας. Προτού μπούμε τώρα στη συζήτηση, θα ήθελα να ζητήσω από τη Φραντσέσκα να προσθέσει και αυτή αν θέλει να πει κάτι σε σχέση με τον τρίλογο. Grazie, Presidente. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμμετείχα στον τριμερή διάλογο ω εισηγήτρια αρμόδια για τον προπολογισμό του 2012, διότι η Κομισιόν πρότεινε στις 21 Μαρτίου να αυξηθεί το επίπεδο των πληρωμών κατά 18 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης για τις πλημμύρες που έγιναν τον περασμένο Οκτώβριο στην Ιταλία, στην Λιγουρία και στην Τοσκάνη. Η Κομισιόν ζήτησε λοιπόν 18 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές έτσι ώστε να μπορούν αυτά τα, τα, τα, κονδύλια να χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το Συμβούλιο είπε ότι το σημειώνει αλλά ότι δεν είχε ακόμα την δυνατότητα να δώσει τη θέση του. Η Κομισιόν ζήτησε να δοθεί γρήγορα λύση γιατί γνωρίζουμε ότι όταν πρόκειται για Ταμείο Αλληλεγγύης ε, είναι πολύ σημαντική η ταχύτητα. Το Ταμείο Αλληλεγγύης που δίνεται μετά από ένα χρόνο αλλιώς ε, γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες. Η Κομισιόν λοιπόν επέμεινε πολύ για την επιτάχυνση. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο όσον αφορά την επιτάχυνση φάνηκε να είναι πολύ πιο διστακτικό. Ο πρόεδρος Λαμασούρ στη διάρκεια της συνάντησης αυτής θύμισε πως πέρυσι είχαμε χρησιμοποιήσει μόνο για αυτό το, ταμείο το μέσο της αρνητικής, του αρνητικού αποθεματικού υπό την Ουγγρική Προεδρία που θα μπορούσε να θεωρηθεί μια λύση επίγουσα για να μπορέσουμε γρήγορα να κινητοποιήσουμε το Ταμείο. Και τώρα περιμένουμε την θέση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει το κατεπήγον σε σχέση, είχε στο παρελθόν ζητήσει το κατεπήγον για το Ταμείο Αλληλεγγύης, αλλά οι καιροί αλλάζουν. Ο Κάλ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Τζοβάνι για την έκθεσή του. About Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα φυσικά ε, οι εξελίξεις που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις, από τις πραγματικές διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό προϋπολογισμό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Δεν υπάρχουν πολλά κονδύλια και έχουμε πολλές ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να έχουμε μια στεναρή, ενισχυμένη και αποφασιστική προσέγγιση, ώστε οι διαπραγματεύσει για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο να διεξαχθούν εκ παραλίλου. Ο σκιώδης μου συγητής, ο κύριος Άλβαρο, σιάζει γιατί βρίσκεται σε αποστολή, του υποσχέθηκα πέραν το θέμα των πληρωμών να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε μόνιμο εισηγητή για τα ΡΑΛ, για τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, τον κύριο Μέλντερ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια καθορίζοντας το επίπεδο πληρωμών που χρειάζονται για να καλύψουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων και αυτό για να διευκαλύνουμε ομαλές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2013. Δεν θα είναι πρώτα πράγματα με το Συμβούλιο, γιατί από ό,τι ξέρουμε οι αντιπροσωπείς στο Συμβούλιο αμφισβητούν την ακρίβεια των αριθμητικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που δεν διευκολύνει μια επικοδομητική συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση πριν περάσουμε στις διπραγματεύσεις. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω γενικά είναι ότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε όπως και πέρυσι ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τα εφαρμοστικά μέτρα για τη στρατηγική του 2020. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2014 για να περιλάβουμε στον προϋπολογισμό μας τις προτεραιότητες τη στρατηγικής του 2020. Θέλουμε ήδη από τον προϋπολογισμό του 2013 να αρχίσουν να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι προτεραιότητες. Ελπίζω να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κάτι άλλο. Πιθανές μεταφορές κονδυλίων για το πρόγραμμα ITER. Ένα θέμα που μάλλον θα ανακύψει εξαιτία τη περσινή συμφωνία, Δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι. Και τέλος, ο σκιώδης ηγετής μας, ο κύριος Άλβαρο, θέλει να εμείνουμε στις δεσμεύσεις μας και τις υποσχέσεις μας για την Παλαιστίνη, γιατί έχουμε συνάψει διεθνείς συμφωνίες. Δεν θα πρέπει να τις αθετήσουμε. Αυτά προς το παρόν, εκ μέρους του σκιώδου ηγετού. Και πιστεύω ότι περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε ενωμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοτμάνης. Thank you very much. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το χειρότερο που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο είναι να διοριστεί γενικό συζητητή για τον προπολογισμό του 2013. <laughs> και θα σα εξηγήσω γιατί το λέω. Έχω και κάποιε προτάσει και ερωτήσει για τον Επίτροπο, τέλο πάντων, τη Γενική Διεύθυνση του Προπολογισμού, τον εκπρόσωπο που έχουμε εδώ. Στην περασμένη συνεδρίαση για κλεισμένο το θηρό με τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι, τι ακούσαμε, ποιο ήταν το βασικό του μήνυμα ότι ήδη το 2012 αρχίζουν κάποια χρηματοοικονομικά τεχνάσματα και κάποια λογιστικά κόλπα, που σημαίνει ότι αν δεν έχουμε χρήματα για να ε, χρηματοδοτήσουμε όλα τα προγράμματα μας, ε, σταματούμε ορισμένα για να πληρώσουμε, βάζουμε από, από το ένα και δίνουμε στο άλλο. Και συνεχώς κάνουμε το ίδιο. Παίρνουμε από τη μια και δίνουμε στην άλλη. Και όταν μας έδωσε το πίνακα με τις χώρες που σταμάτησαν την απορρόφηση των κονδυλίων και ήταν χρωματικό, ε, μας έδειξε και άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία που απορροφούσαν κονδύλια και δεν ήταν κόκκινες. Και μάλιστα μέχρι 50 δισεκατομμύρια, γιατί αυτές οι δύο χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, φοβόνταν ότι θα έχαναν τα κονδύλια. Συνήθως όπως είπε και ο κύριος Λεβαντόσκη, το Δεκέμβριο κρίνονται αυτά, αλλά είμαι σίγουρη ότι ήδη δεν έχουν αρκετά κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν όλα τα προγράμματα. Οπότε, αν αυτό το παρατηρήσαμε ήδη από το 2012, ούτε καν για το 2013, φαίνεται ότι χωρίς διορθωτικούς προϋπολογισμούς δεν πρόκειται ε, να ανεχθούμε τέτοια επικίνδυνα λογιστικά κόλπα γιατί θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και οι χώρες αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Και το 2013 φαίνεται ότι θα είναι δεκαπλάσια ανάγκη για τέτοια λογιστικά τεχνάσματα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ε, σε όλες τις δημοσιονομικές προοπτικές και στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, τα περισσότερα κονδύλια που δόθηκαν για πληρωμές και αναλήψεις υποχρεώσεων αφορούσαν τη συνοχή. Δεν ξέρω γιατί οι αναλήψεις υποχρεώσεων ήταν ε, ισότιμα κατανεμημένες. Ε, ε, ένα έβδομο κάθε χρόνο για την επταετία των δημοσιονομικών προοπτικών. Και ξέραμε ότι οι πληρωμές των ε, πρώτων δύο χρονών ήταν μηδενικές, οπότε κανονικά οι πληρωμές ήταν μηδενικές, όπως ε, έγινε τελικά το 2007 και το 2008 είχαμε μόνο προκαταβολές, που ήταν ουσιαστικά μόνο 10% των αναγκών. Αυτό σημαίνει ότι η αναλήψη υποχρεώσεων από χώρες, ε, ε, στις χώρες για την πρώτη διετία δεν χρησιμοποιήθηκαν, οπότε θα τις ζητήσουν αργότερα, το 2012-2013, πολύ περισσότερο από το 1 έβδομο που κανονικά είναι η ισότιμη κατανομή στην επταετία. Και έχουμε το δεύτερο πρόβλημα που κάνει ακόμη πιο δύσκολη αυτή την λογιστική ε, κατανομή και τα τεχνάσματα αυτά. Είχαμε ε, το 2009 τις άλλες δραστηριότητες και χρησιμοποίησαμε τα κονδύλια. Είχαμε καταρχήν το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης 5,6 δισεκατομμύρια, 1,2 ε, είχαμε οικονομίες και αν προσθέσουμε και κάπου, κάποια κονδύλια αριστερά και δεξιά έχουμε 2 δισεκατομμύρια αυτά τα κονδύλια δόθηκαν στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Οπότε η εκπλήρωση των υποχρεώσεων δεν θα αφορά του στόχου τη συνοχής, αλλά άλλου σκοπού. Και φτάνουμε στο πολιωτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2012-2013. Και πού πάνε αυτά τα χρήματα? Έχουν κάνει φτερά. Οπότε, αν η αρχική κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν επταετή προπολογισμό με συγκεκριμένη κατανομή και ορισμένα κονδύλια χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο, δεν πρόκειται να δοθούν συμπληρωματικά κονδύλια. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, χρειαζόμαστε ομοφωνία στο Συμβούλιο και ενισχυμένη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Οπότε, ερωτώ τον εισηγητή τι θα γίνει το 2012 και το 2013. Και ρωτάμε και τις γενικές διευθύνσεις ε, προπολογισμών και περιφερειακής ανάπτυξης. Από πού θα βρουν τα χρήματα για να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το 2012 και 2013 και τις πληρωμές για αυτά τα δύο χρόνια που θα είναι πολύ ε, περισσότερες από τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τα RAL, τα LIQUIDE, τα υπόλοιπα προς εκαθάριση. Από νομική άποψη είναι δεμένα τα χέρια μας, γιατί ε, από το παράδειγμα της 5 το Δεκέμβριου βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ε, διέξοδος. Γιατί φτάνουν οι λογαριασμοί και πρέπει να πληρωθούν. Οπότε μένουν τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, που λέει ο, Λε, Λεβαντόσκι είναι 207 και λίγο παραπάνω εκατομμύρια. Είναι αποθεματικό. Ότι ε, αυτά που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει είναι αποθεματικό. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε για την επτέτεια. Πραγματικά, ε, δεν ξέρω τι απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντω, αν υπήρχαν υποχρεώσει, αναλήψεις υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμέ τη ε, συνοχή. αλλά ε, εν μέσω τη κρίση με πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δοθούν για άλλου σκοπού. τότε πώ θα καλυφθούν τα προγράμματα τη συνοχή? Η μόνη απάντηση που θα μπορούσε νομικά τουλάχιστον να μα δώσει η νομική επιτροπή είναι ότι όλε οι πληρωμές που έγιναν για άλλου σκοπού έχουν ε, εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οπότε την ευθύνη τη μοιράζονται και τα τρία θεσμικά όργανα. Αλλά αυτά όμως δεν αλλάζουν την αριθμητική κατανομή στην επταετία. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον εισηγητή, όχι μόνο για το 2013, αλλά και για το 2012. Γιατί θα έχουμε προβλήματα, όχι σε αρχές του χρόνου. Έχουμε πρόβλημα με την όλη φιλοσοφία των δημοσιονομικών προοπτικών. Μπορούμε να αλλάξουμε την νομοθεσία για να χρησιμοποιούμε τα αρέστα ελικίντα, τα ραλ και όταν ε, δεν ε, ε, χρησιμοποιούνται κάποια κονδύλια να τα κόβουμε και να τα δίνουμε αλλού ή αν πάμε σε διορθωτικό προπολογισμό πότε θα φτάσουμε στα ανώτατα όρια και μπορεί να τα ξεπεράσουμε και αυτό θα είναι δύσκολο. Μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως με βάση τα στοιχεία έχω προβληματισμούς και ερωτήσεις και απαντήσεις δεν βρίσκω. Και δεν ξέρω τι θα γίνει στο τριήμερη διάλογο, στη συνδιαλλαγή. Εκεί θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα ερωτήματα από αυτά που μας έθεσε πριν από λίγο η συγγετής. Βεβαίως. Το θέμα της ε, δημοσιονομικής μηχανικής της Κομισιόν μέσα σε εισαγωγικά δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει αδιάφορος. Όταν τελειώσουμε αυτό το γύρο θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και ίσως μπορούμε να πάρουμε την Κομισιόν μια πρώτη δόση ε, απαντήσεων. Εγκαρία Ζαβάλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Γιώτα. Εμείς βλέπουμε πολύ θετικά και πολύ αισιόδοξα αυτή την κατάσταση ως αποτέλεσμα αυτής της ε, συνάντησης που φυσικά δεν ήταν διάλογος ούτε τριάλογος αλλά μονόλογος αλλά προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα θετικά. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι με αυτή τη συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο τουλάχιστον έχουμε τα ίδια αριθμητικά στοιχεία για τα οποία μπορούμε να εργαστούμε για τη συνδιαλλαγή και δεν γίνεται αυτό που έγινε στο παρελθόν να παίζουμε με άλλες τράπουλες και επίσης τουλάχιστον το Συμβούλιο αποφάσισε και αποδέχτηκε ότι πρέπει να εξισορροπήσει κάπω τα μέτρα λιτότητα με τι απαραίτητε πολιτικέ ανάπτυξη. Αυτό μα κάνει κάπω πιο αισιόδοξου, αλλά πιστεύω ότι η θέση που κατέδειξε το Συμβούλιο στην πρόσφατη αυτή συνάντηση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Γιατί αυτό το οποίο λέει το Συμβούλιο είναι πρέπει να αφήσουμε ένα επαρκές περιθώριο για τον προπολογισμό του 2013 μέχρι τα όρια των δημοσιονομικών ε, προοπτικών και αυτό το οποίο θέλει να κάνει το Συμβούλιο, αν τα ερμηνεύσω σωστά, είναι όχι να είναι ρεαλιστικό, αλλά να μειώσει τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Αν ξεκινήσουμε από ένα σχετικά μικρό προϋπολογισμό, περιορίσουμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων και χρειαζόμαστε να βρούμε από κάπου αλλού 360 εκατομμύρια για το ίτερ και συγχρόνως έχουμε και την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας μένει ελάχιστο περιθώριο λοιπόν, Δεν ξέρουμε από πού θα βρουν χρήματα για να υποστηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν τις πολιτικές αυτές που λένε ότι θα αντισταθμίσουν τις πολιτικές λιτότητες στα κράτη-μέλη. <clears throat> Όπως είπε και ο κ. Κοτσμάνης, δεν είναι εύκολο να, δεν είναι εύκολο να είναι κανείς εισηγητής και σίγουρα δεν είναι εύκολο για κανένα από εμάς να αντιμετωπίσουμε τον προϋπολογισμό του 2013. Θα πρέπει να κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα, όλες τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο. Και αν ήταν δύσκολα τα πράγματα στο παρελθόν, τώρα εφέτος είναι ακόμα πιο δύσκολο και θα είναι γυρίζει, η βίδα γυρίζει ένα γύρο παραπάνω και μας πιέζει λίγο περισσότερο. Θα είναι λοιπόν δύσκολη αυτή η διαπραγμάτευση και θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ο παράγον του δημοσιονομικού πλαισίου από το 2014 που θα μπερδέψει ακόμα περισσότερο τη συζήτηση. Εμείς πάντως πρέπει να μείνουμε στη θέση μας και να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τον προϋπολογισμό, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα περιθώρια της ευελιξίας για να χρηματοδοτήσουμε το ίτερ και φυσικά η είσοδος της Κροατίας <clears throat> θα πρέπει να οδηγήσει σε τροποποίηση του χρηματοδοτικού πλαισίου, του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως έγινε με οποιαδήποτε ένταξη νέας χώρας στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη και από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Όταν λέει το Συμβούλιο ότι θέλει να συνενώσει κάποιες πιστώσεις υποχρεώσεων, να τις ε, συγχωνεύσει. Αλλά το θέμα είναι πού θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε μια συγχώνευση. Γιατί η κάθε πίστοση υποχρεώσεων έχει μια βάση. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε εφεύρει. Είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα συμφωνίας και με το Συμβούλιο θεμητές προσδοκίες σε σχέση με όλα αυτά τα κονδύλια που μπορούν να οδηγήσουν και σε προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ δεν θέλω να αντιμετωπίσω μια κατάσταση <clears throat> όπου ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν είναι εύκολο το έργο του Τζοβάνι λοιπόν. <clears throat> Θα πρέπει όμως όλοι να τον βοηθήσουμε και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε σαφές αυτό και προς το Συμβούλιο ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Ο Ευχαριστώ. Για το θέμα αυτό, νομίζω ότι φαίνεται ότι το μόνο θεσμικό όργανο που πραγματικά ενδιαφέρεται για τα κράτη-μέλη είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όταν μιλούμε για πιστώσει πληρωμών, μιλούμε για πιστώσει πληρωμών των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να αναλάβουν τι ευθύνε του και τι υποχρεώσει του. Κάτι που είναι προ το δικό του συμφέρον τελικά και υποσκάπτουν την ίδια του τη θέση. Μόνο εμείς ενδιαφερόμαστε για τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο φαίνεται ότι στρέφεται κατά του εαυτού του. Τα θεσμικά όργανα πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και ως προς τις ε, υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, αλλά και απέναντι στους πολίτες. Και αυτή είναι η λέξη κλειδί, η αξιοπιστία. Οι υποχρεώσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο, οι δεσμεύσεις για τις πληρωμές, θα πρέπει ε, να τηρηθούν, να τη στηρίσει. Και ε, περνάμε στο Ταμείο της Ελληνικής. Το Ταμείο Ελληνικής έχει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Το ίδιο το Συμβούλιο ανέλαβε τη δέσμευση και με σχετικό κανονισμό ότι θα είναι ένα ταμείο που θα κινητοποιείται, θα ενεργοποιείται γρήγορα και θα καλύπτει έκτακτες ανάγκες. Γιατί λοιπόν καθυστερεί τη διαδικασία αυτή. Γιατί κολλησιέργει το Συμβούλιο, παρόλο που το ίδιο συμφώνησε να καλύπτει κατεπίγουσες ανάγκες, ό,τι αφορά την Ιταλία για το δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό για την Τοσκανία. Ε, αυτό, ανέφερε το, αυτό αναφερόταν στον Οκτώβριο του 2011. Και μίλησαμε για ζημιέ 722 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η πρόταση αφορά 18 εκατομμύρια ευρώ. Αν το Συμβούλιο που έχει εγκρίνει το κανονισμό και που έχει ένα δισεκατομμύριο Ταμείο Λεγγύης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δίνει μόνο 18 εκατομμύρια. Οπότε, προς τι αυτό το Ταμείο Λεγγύης, γιατί το δημιουργήσαμε, αν το ίδιο το Συμβούλιο λέει ότι θέλει να αναστείλει τη λειτουργία του. Γιατί τα 18 εκατομμύρια είναι μόνο 2,5% του συνόλου των ζημιών. Και αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο της, χρηματο... της αλληλεγγύης δεν πρέπει να καθυστερεί ούτε να παρεμποδίζεται. Θα πρέπει το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν να αναλάβει τις ευθύνες του, να δείξει την φερέγγια συμπεριφορά του και όταν αναλαμβάνει δεσμεύσεις να τις στηρεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Τζοβάνι για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, γιατί και επίσης γιατί καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι το έργο του εισηγητή για τον επόμενο προπολογισμό. Αλλά πιστεύω πως ο εισηγητή του επόμενου προπολογισμού θα είναι αξιόπιστο στο βαθμό που αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα του δώσουν την ισχύ για να μπορέσει να διαπραγματευτεί. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι χωρί τα κατάλληλα κονδύλια όσον αφορά τις ε, ε, πιστώσεις πληρωμών, το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα είναι αξιόπιστο και ο προϋπολογισμός δεν θα είναι εφαρμόσιμος ε, εκτελέσιμος. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μαζί ε, στη διάρκεια της ε, διαδικασίας ακολουθώντας αυτή την έλεγχο που ανέλαβε να κάνει η Κομισιόν και να μας ενημερώνει γιατί πώς προοδεύει οι διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι ανάγκες για τις Επιστώσει πληρωμών. Πιθανότατα θα πρέπει να κάνουμε θαρα, ε, θαραλές επιλογές και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί γιατί πολλοί συνάδελφοι ε, παρενέβησαν προ αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα δώσει ισχύ στον εισηγητή και κυρίω αξιοπιστία στο θεσμικό μας όργανο. Επιπλέον, ε, μάλλον με άλλα λόγια, θα πρέπει Καθώ η διαδικασία είναι μόλις στην αρχή, γιατί ο εαρινός τριμερή διάλογο είναι μόνο μια πρώτη επαφή όπου αποφασίζεται το χρονοδιάγραμμα και ο καθένας παρουσιάζει τις προτεραιότητές του. Εμείς στις κατευθύνες γραμμές για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου εξ αρχής δώσαμε σημασία στις, στα θέματα των πληρωμών γιατί είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ώστε ο προπολογισμό να μπορεί να εκτελεστεί. Γιατί το δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να κλείσει. Αν τώρα είχαμε αναλάβει υποχρεώσει που στενά συνδέονται με νομικέ βάσει, είναι προφανέ ότι θα πρέπει αυτέ οι υποχρεώσει να πληρωθούν. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκοτμάνης, σαφώς η πολιτική συνοχή μέχρι στιγμή, περιλάμβανε πολλές υποχρεώσεις, γιατί αυτό είναι συνειφασμένο με την ίδια στην ε, πολιτική, γιατί είναι ιδιαίτερα για τις υποδομές. Υπάρχει μια περίοδος υποχρεώσεων και μετά ακολουθούν οι πληρωμές. Αυτό, ναι, διευρύνει το ράλο, αλλά στο τέλος του δημοσιονομικού πλαισίου όλα αυτά ε, μεταφέρονται σε ένα πλαίσιο λειτουργικότητας των, προγράμμα, των προγραμμάτων και γι' αυτό και χρειάζονται οπωσδήποτε να γίνουν οι πληρωμές. Θα κλείσω με ένα στοιχείο που εμείς ε, ανέκαθεν τονίζαμε, αλλά φέτος το βάλαμε και στις κατευθυντήριες γραμμές και το υπογραμμίσαμε και στο Συμβούλιο, ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι στα τελευταία δύο χρόνια στην, συνδιαλλαγή παρουσιάστηκε ορίζοντας ένα μάξιμο με επίπεδο των περικοπών των πληρωμών, χωρίς να λέει πού θα πρέπει να γίνουν αυτές οι περικοπές. Ωραία λοιπόν. Αν το Συμβούλιο θέλει να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, να αναλάβει και την ευθύνη αυτή τη πορεία που θέλει να ακολουθήσει. Η πολιτική συνοχή, όπω είπαν σωστά οι συνάδελφοι, είναι στο κάτω-κάτω λογαριασμοί που τελικά επιστρέφουν στα κράτη-μέλη. Και άρα το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι στην ουσία οπλίζει μια γροθιά που θα το χτυπήσει το ίδιο στο, στο πρόσωπο. Το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο παρακολουθεί και προσέχει αυτή τη βούληση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ώστε να διατηρηθεί δραστήρια και αποτελεσματική η πολιτική συνοχή. Εάν η Κομισιόν στο τέλος του ε, 11. με τα λιγοστά κονδύλια που είχε στο ταμείο της θέρισε να ε, καθαρίσει κάποιες χώρες όπως αυτές που είπε ο συνάδελφος Γκοντμάνης που ήταν η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες ρευστότητας αυτό δεν μπορεί να σταθεί για πολύ καιρό, ούτε να συνεχίζεται για πολύ καιρό. Και είναι σαφέ ότι πρέπει εδώ να ενεργήσουμε στεναρά στη στρατηγική μα στο πλαίσιο του 2013, δείχνοντα ε, δείχνοντας ε, τις δυνάμεις μας και ακόμα και χτυπώντας τη γροθιά μας στο τραπέζι. Μερσή, λέει πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο, στη δεύτερο τμήμα του ιταλικού μου ντουέτου, τη, τη Φραντσέσκα. Ε, Όπως είπε ο συνάδελφος Φερνάντες, για το ε, Ταμείο Αλληλεγγύης φυσικά και διακυβεύεται η αξιοπιστία μας και η αξιοπιστία αυτού του κοινοβούλιο, αν και συχνά Όντω τα κονδύλια είναι πολύ μικρά σε σχέση με τι ζημιέ που υπέστησαν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει τώρα να δούμε πώ θα αντιδράσει συγκεκριμένα το Συμβούλιο. Και μετά θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τη δική μας θέση ως Κοινοβούλιο και που όπως είπα και στον τριμερή διάλογο είναι πλήρη στήριξη στην θέση τη ε, Κομισιόν που είναι πιο ξεκάθαρη γιατί είπε ότι πρέπει όντως να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να βρούμε και ειδικέ τεχνικές για να μπορούμε να εκταμιεύσουμε γρήγορα αυτά τα κονδύλια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου που όπως σας είπα φάνηκε πιο διστακτικό και προσεκτικό αυτή την πρώτη φάση. Ευχαριστώ Φραντσέσκα. ο Γενικός Διευθυντής της Κομισιόν τώρα για να κλείσει το σημείο 4 και αν μπορεί να μας δώσει ίσως και κάποια απάντηση στο ερώτημα του κύριου Γκοτμάνης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όταν αναφέρθηκε σε δημοσιονομική σε έργα δημοσιονομικού μηχανικού μάλλον ο κύριος Λεβαντόφσκι χρησιμοποίησε μία εικόνα που για ορισμένου σημαίνει ζογκλερισμό οικονομικό, δημοσιονομικό <clears throat> για να αντιμετωπιστούν σημαντικές πιστώσεις πληρωμών οι οποίες ήταν υπερβαίνουσες αυτών των ποσών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες ουσιαστικά εμφανίστηκαν στο Δεκέμβριο του 2011. Ξέρετε ότι εμείς τηρώντας πάντα τους κανόνες έχουμε ένα περιθώριο δύο μηνών για να εκτελέσουμε αυτές τις πληρωμές. Η αρχή του χρόνου είναι πάντα δύσκολη γιατί θα πρέπει να πληρώσουμε, να δώσουμε πίσω στα κρατημέλη τις άμεσες επιδοτήσεις που έχουν καταβάλει στον αγροτικό τομέα. Στο σύνηθες λοιπόν βάρος εργασίας προσθέθηκε και ένα πρόσθετο άχθος που αφορούσε <clears throat> αυτό το ποσό των 5 δισεκατομμύριων ευρώ που έπρεπε να καταβληθεί μετά από την απόφαση του Δεκεμβρίου. Εμείς ξεκινήσαμε με το να αντιμετωπίσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την σωστή διαχείριση των ποσών που είχαμε στο ταμείο μας, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των προθεσμιών. Περάσαμε αυτή την ερημική χρονική περίοδο και ίσως κάπως καθυστερήσαμε για ορισμένε πληρωμές, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στις αρχές Απριλίου όλες οι πληρωμές, μα όλες οι πληρωμές, οι οποίες για τις οποίες είχε γίνει εντολή προς την Κομισιόν να πληρωθούν και μέσα στα πλαίσια της ευθέτου τάξης όλες αυτές οι πληρωμές θα έχουν γίνει μέχρι τον Απρίλιο. Επομένως εμείς θα έχουμε διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη φάση επιτυχώς και στις αρχές Απριλίου δεν θα υπάρχει ούτε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν θα έχει λάβει τα ποσά τα οποία πρέπει να του καταβληθούν επί τη βάση των στόχων που είχαμε να καταβάλουμε εμπρόθεσμα όλα αυτά τα κονδύλια στα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια των διαθεσιμοτήτων του προϋπολογισμού. Τώρα κάτι διαφορετικό είναι αυτό το οποίο θα γίνει στο δεύτερο μέρος του έτους. Η εμπειρία του τέλους του 2011 καταδεικνύει ότι δεν αποκλείεται και πάλι να παρουσιαστεί μια ισχυρή πίεση σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών η οποία θα συσσωρευτεί κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο τμήμα του έτους. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, <clears throat> μια πιθανότητα που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, ότι πράγματι μπορεί να βρεθούμε στα στενά σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών τότε η Κομισιόν θα υπομειστεί τις ευθύνες της και θα διαχειριστεί αυτά τα κονδύλια όπως οφείλει να πράξει κάτω από τέτοιες συνθήκες, έχοντας πάντα κατά νου την δήλωση η οποία έχει διατυπωθεί και εγκριθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2012 σε ό,τι αφορά το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών. Αλλά θα σας πω κάθε πράγμα στον καιρό του. Υπάρχουν πολλές τεχνικές του προϋπολογισμού που είναι γνωστές και μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τις εντάσεις σε σχέση με τις απαιτούμενες πληρωμές. Υπάρχουν μεταφορές πιστώσεων. Και όταν αυτό είναι απαραίτητο προτείνουμε μεταφορές πιστώσεων και αν αυτό είναι δυνατό μπορούμε να προχωρήσουμε όπως προσπαθήσαμε ήδη να κάνουμε πέρσι με αποτελέσματα τα οποία ήταν περιορισμένα. Μιλούσαμε για 500 εκατομμύρια ευρώ και αυτό έτυχε ε, έγκριση και στην πραγματικότητα ήταν πολύ λιγότερα τα ποσά τα οποία απαιτήθησαν. Αυτό το οποίο είναι στο τέλος του 2012 ήταν ότι μια σειρά από κράτη-μέλη εξέφρασαν τη θέλησή τους να τους καταβληθούν ορισμένες πληρωμές για να μην είναι θύματα του κανόνα που ακυρώνει κάποια κονδύλια. Το νησιν 3 παραδείγματο χάρη. Εφέτο θα υπάρξουν πάλι αντίστοιχε πιέσει. Αλλά προ το παρόν δεν ξέρουμε ακριβώ σε τι ύψο θα είναι τα κονδύλια αυτά τα οποία θα απαιτηθούν. Προηγουμένω ετέθηκε κάποια αμφιβολία σε σχέση με τι στατιστικέ τη Κομισιόν τα στοιχεία τα οποία σας δίνουμε και σε εσά και στο Συμβούλιο παραλλήλως είναι σοβαρά στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία καθορίζονται επί τη βάση των πληροφοριών που μας δίδονται σε σχέση με την επιμερισμένη διαχείριση από τα κράτη-μέλη. Και κατανοείται ότι για ό,τι δεν είναι στην επιμερισμένη διαχείριση και τα διαχείριζεται μόνο η Κομισιόν, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Αυτά μπορώ να σας πω λοιπόν σε σχέση με την αρχή του έτους αυτού και το θέμα των ταμιακών αποθεμάτων μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων πληρωμών για το υπόλοιπο τμήμα του έτους και τέλος <clears throat> σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2013 νομίζω ότι ο Επίτροπος Λεβεντόφσκι έχει ήδη εκφράσει την άποψή του με μεγάλη σαφήνεια και η Κομισιόν θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα παρουσιάσει μια ρεαλιστική πρόταση. Δηλαδή μια πρόταση η οποία εδράζεται επί αυτών τα οποία θα μπορούμε ευλόγως να αναμένουμε σε ό,τι αφορά τις αιτήσει πληρωμών για το 2013, το οποίο είναι το ίστατο έτος της τωρινής δημοσιονομικής περίοδου, όπως υπενθύμησαν πολλοί βουλευτές. Αυτά μπορώ να σας πω λοιπόν υπό μορφή απαντήσεων και σχολείων σε αυτά που είπε ο κύριος Γκοτμάνης. Σας ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι οι προοπτικές για τις διαπραγματεύσεις και ο χρόνος που μας μένει για αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν είναι πολύ άνετος. Και οι προοπτικές δεν είναι πολύ άνετες. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο τώρα Έχουμε τώρα την έκθεση για το διορθωτικό προϋπολογισμό για, για, το, για τους ίδιους πόρους και θα ήθελα εδώ να παρακαλέσω να δώσετε μία σύντομη παρουσίαση short report. On the contact group or on the... On the GAC and the contact group. You can do it all together. It speeds up. Thank you, Madam Chair. basically... Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, τρία πράγματα έγιναν. Θα είμαι πολύ σημαντικό. Θα είμαι πολύ σύντομος από τη διάσκεψη για του ίδιου πόρου και το πολιτέ δημονομικό πλαίσιο. Νομίζω πολύ πήρα, πήρα μέρος και παρακολουθήσαμε τη διάσκεψη. Πολύ καλό φόρουμ, ε, πολύ καλές παρουσιάσεις ε, μεταξύ άλλων του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και νομίζω ότι όλοι όσοι έλαβαν μέρος και παρακολούθησαν ε, συμφωνούν ότι μπορεί να μην Υπήρξε ομοφωνία, αλλά η συζήτηση ήταν επικοδομητική και ακούστηκαν πολλά επιχειρήματα. Όλοι είχαν ε, τα επιχειρήματά τους ε, και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για τη συζήτηση. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους για να επικοινωνήσουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε ό,τι αφορά το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Δευτέρας. Ο συνήθως μας ενημέρωσαν και πριν και μετά το Συμβούλιο το, Συμβούλιο αυτό εξέτασε το πρώτο πακέτο της ε, Δημοσιονομικής Συμφωνίας που θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τον Ιούνιο και αυτό το πακέτο δεν περιλαμβάνει τα δύο πιο σημαντικά θέματα, την συνοχή και την κοινή γεωργική πολιτική. Η Προεδρία υπέβαλε ένα έγγραφο που υπέβαλε και στα κράτη-μέλη, έγινε συζήτηση, αλλά δεν είναι σαφές ακόμη για ποια σημεία υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή αν θα αποκρισταλωθεί μια ενιαία θέση στο Συμβούλιο. Πάντως πολλά ζητήματα εξετάστηκαν που είναι σημαντικά και για μας. Το πρώτο αφορά ένα ζήτημα αρχής για μας που αφορά και τον τρόπο οργάνωση των εργασιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα προβλήματα και τα ζητήματα που περιλαμβάνει το διαπραγματευτικό πακέτο. Γιατί έχουμε δύο διαδικασίες. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το διάλογο δηλαδή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το ίδιο το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ε, τη νομική βάση που είναι η συναπόφαση. Ενώ στο πρώτο θέμα έχουμε άλλη νομική βάση και υπάρχει μια σύγχυση πολλές φορές για το ποια διαδικασία θα εφαρμόσουμε για να λύσουμε τα προβλήματα. Το επόμενο θέμα θα είναι συνοχή και γεωργική πολιτική. Και φαντάζομαι οι συνάδελφοί μας σε άλλες επιτροπές ε, θα προσέξουν ιδιαίτερα τα ζητήματα που θα μπουν στην πολιτι... στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και έχουμε και το θέμα της νομικής βάσης ε, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτά είναι τα γενικά σχόλια. Πάντως, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολος ο διαχωρισμός των θεμάτων. Δεν είναι σαφές τι περιλαμβάνονται στα τομεακά ζητήματα και τι στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο συμβούλιο, Έγινε απευθεία αναμετάδοση των εργασιών, οπότε όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειε μπορούν να το παρακολουθήσουν στο ίντερνετ. Κάποιες χώρες μίλησαν για το γενικό όγκο του προϋπολογισμού, ζητώντας περικοπές σε όλα τα κεφάλαια, σε όλους τους τίτλους. Και φυσικά Γνωρίζουμε τους συνήθεις υπόπτους, τις 8 χώρες δηλαδή που υπέγραψαν μια επιστολή σχετικά. Έγινε συζήτηση και για την ελαστικότητα, την ευελιξία, άλλο σημαντικό ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Μιλάει για ελάχιστη ελαστικότητα των, των προϋπολογισμών ελάχιστο περιθώριο, λίγο κάτω από το ανατοτόριο, ενώ, ενώ μερικές χώρες του μεγαλύτερη ελαστικότητα και άλλες μικρότερη ελαστικότητα. Υπάρχει και μεταξύ των κρατών μελών διάσταση απόψεων. Μερικές χώρες δεν θέλουν κανένα απόλυτο περιθώριο λιγμών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητήσεις έγιναν για το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο θα πρέπει να είναι εντός ή εκτός ε, του προπολογισμού. και για τη χρηματοδότηση του GMES. Εμείς είπαμε να είναι εντός του προπολογισμού, αλλά με αντίστοιχα ανώτατα όρια και τα απαραίτητα κονδύλια. Και για το θέμα αυτό υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα, για τα κατά πόσο εν ώψη του 2020 θα πρημοδοτείται, θα χρηματοδοτείται μόνο η επιστημονική αριστεία ή και μια πορεία προς την επιστημονική αριστεία, δηλαδή και οι επιστημονικές βάσεις που θα αναπτύσσονται από κάποιες χώρες μέλη. Δεν θα επιμείνω στα θέματα αυτά. Αν σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως, κοιτάξτε στο ίντερνετ. Κάθε χώρα έχει τρία λεπτά για να υποστηρίξει τη θέση της. Η Προεδρία έμεινε ικανοποιημένη από τη συζήτηση, είπε ότι ήταν αρκετά ήρεμη. Θα δούμε ποια θα είναι τελικά η έκβαση της συζήτησης. Το επόμενο, το επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα γίνει τον Απρίλιο στο Λουξεμβούργο και θα ασχοληθεί με τη συνοχή και την κοινή γεωργική πολιτική. Προς το παρόν πάντως η Προεδρία τηρεί το χρονοδιάγραμμα που είχε θεσπίσει. Το Μάιο θα προσπαθήσει να θέσει σε συζήτηση το ενοποιημένο έγγραφο, χωρίς όμως τα στοιχεία του διαπραγματευτικού πακέτου και κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο θα το υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο. Αυτά για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Τώρα, δύο λόγια για την ομάδα επαφής που συνεδρίασε την εβδομάδα αυτή. Ένα από τα βασικά θέματα που έθεσε ο πρόεδρος Σούλτ στην ομάδα επαφή είναι και πάλι η εσωτερική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις, εξε... συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δύο σημαντικά ζητήματα έχουμε εδώ. Πρώτον, σε τι στάδιο θα πρέπει οι επιτροπές να εφαρμόζουν την αρχή ότι αν δεν συμφωνηθούν όλα, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Δηλαδή, να αποφεύγεται συμφωνία για κατακαιρματισμένα τμήματα, για μερικά μόνο τμήματα. Πάντως, η ομάδα επαφή συμφώνησε να ε, ζητήσει ο πρόεδρο Σούλτ από του πρόεδρου τη Επιτροπή να σταματάνε πριν την πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή, η συζήτηση για την νομική βάση να παραμένει σε επίπεδο Επιτροπή. Θα φαντάζεστε ότι κάποιοι πρόεδροι επιτροπών θα ήταν πιο φιλόδοξη. Αλλά προς το παρόν η λύση αυτή επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εφαρμόσει μια πιο ενιαία διαδικασία και πιο πάγια. Τέλος, στην προηγούμενη συνεδρίαση της ομάδας επαφής, πολλοί ε, πρόεδροι επιτροπών ζήτησαν χρονοδιάγραμμα, ένα χρονικό ορίζοντα. Υπάρχει αυτή η πρόταση ήδη. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου το συζήτησε και με τον πρόεδρο Λαμασούρ και έχουμε πια ένα προτινόμενο χρονοδιάγραμμα, ιδιαίτερα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και με την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε, θα αναφέρω μερικά ορόσημα. Θέλουμε πάντως να έχουμε μια ενδιάμεση έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο, αφού αποκρισταλωθεί, οριστικοποιηθεί η, η θέση του Συμβουλίου για το διαπραγματευτικό πακέτο που θα έχουμε το διαπραγματευτικό πακέτο τον Ιούνιο ή Ιούλιο, θα γίνει συζήτηση στις ειδικέ επιτροπές, θα ψηφίσουν τις γνωμοδοτήσεις τους τον Σεπτέμβριο και αρχές Σεπτεμβρίου, 6 Σεπτεμβρίου, στην Επιτροπή μας θα έχουμε την πρώτη συζήτηση του σχεδίου ενδιάμεσης έκθεση προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τη διαδικασία στις αρχές Νοεμβρίου. Οπότε να αντιδράσουμε εγκαίρως και πριν το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στη θέση του Συμβουλίου. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλο σωστό αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ίσως χρειαστεί να εγκρίνουμε κάποιο ψήφισμα το Μάιο πριν το Συμβούλιο του Ιουνίου για να δώσουμε κάποιες κάποια μηνύματα εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι βέβαιο ακόμη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και αν παραστεί ανάγκη να στείλουμε πιο ηχηρά μηνύματα πριν το Συμβούλιο τη διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου, θα το κάνουμε μέσω ψηφίσματο. Αλλά αυτό θα αποφασιστεί αργότερα. Αυτά για το τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει δώσει, θα δώσει μάλλον τις πληροφορίες αυτές και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όλοι οι συνάδελφοι στις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να πράξουν τα απαραίτητα ώστε επί τη βάση των νομοθετικών αυτών αποφάσεων να συνεχίσουν την εργασία τους. Δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν είναι ότι θα πρέπει να τα παγώσουμε όλα μέχρι το καλοκαίρι μέχρι το μετά από τις διακοπές. Συνεχίζεται η επεξεργασία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και είναι απαραίτητο αυτό να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για τις αρχές και τις απαραίτητες κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των επιμέρους πολιτικών. Να υπάρξει συζήτηση και διαμόρφωση κοινή θέση. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο σε σχέση με αυτό το σημείο. Όχι, δεν βλέπω κανένα να το θέλει. Α, ο κύριος Ρικέ. Ουφ. Ένα ερώτημα μονάχα λέει ο κύριος Ρικέ. Νομίζω ότι έχουμε μία αναδυόμενη ε, συνένεση στο ότι οι επιτροπές δεν μπορούν να εργαστούν επί συγκεκριμένων αριθμητικών ποσών. Μπορούμε να μιλήσουμε για κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να ψηφίσουν επίσημα οι επιτροπές τα ψηφίσματά τους τα αντίστοιχα χωρίς αριθμούς και θα πρέπει να επανέλθουμε για δεύτερη φορά ε, με συγκεκριμένους αριθμούς ή θα κλείσουμε την ε, νομοθετική επεξεργασία χωρίς να ψηφίσουμε και θα περιμένουμε να έρθουν τα αριθμητικά στοιχεία. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει οι επιτροπές να γνωρίζουν ποια είναι η θέση της Επιτροπής Προϋπολογισμών στο θέμα αυτό για να ξέρουν διαδικαστικά πότε θα ψηφίσουν, αν θα ψηφίσουν με αριθμού ή αν θα ψηφίσουν αργότερα μονάχα του αριθμού. <clears throat> Αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί και ο πρόεδρος Σούλτς θα το ελέξει πάλι με την ε, συνέλευση των Προέδρων σε μια έκκληση που θέλει να κάνει για αυτό το πράγμα. Όλες οι επιτροπές θα φτάσουν στο τέλος της εργασίας τους χωρίς στοιχεία και δεν θα έρθουν οι εκθέσεις τους στο, στην Ολομέλεια. Θα έρθουν στην Ολομέλεια μόνο όταν έχει υπερατωθεί η διαδικασία και θα έχουμε τους αριθμούς. Επομένως, επεξεργασία στο εσωτερικό κάθε επιτροπής, χωρίς στοιχεία και χωρίς να φτάσουν στην Ολομέλεια. Επομένως, τυπικά δεν κάνουν την ε, επεξεργασία αυτή. Μόνο στην Επιτροπή. Θα ψηφιστούν στην Επιτροπή χωρίς αριθμούς οι θέσεις τους. Όλα γίνονται όλα γίνονται, όλα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε και για ποσοστά παραδειγματο χάρη. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι όλες οι βασικές αρχές θα πρέπει να έχουν γίνει σαφείς στις επιτροπές και θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση όταν έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας. αυτό που είπε ο Ντομινίκ είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο Σαλβαδόρ, γιατί είναι και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών ο κύριος ε, Ρικέ. Αν πρέπει να κάνει Επιτροπή Μεταφορών σε σχέση με το Connecting Europe Facility, Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσει παραγωγή το όριο αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν, αν ψηφίσει την νομοθετική αυτή ε, έκθεση θα πρέπει να έχει στοιχεία τα οποία είναι αξιόπιστα. Είναι πιο εύκολο να φέρουμε τελικά τις ε, τελικές αποφάσεις στην ολομέλεια και να μείνουμε στις επιτροπές σε επίπεδο γενικό. Είναι διαφορετικό το θέμα για τα θέματα συνοχής και για τα θέματα γεωργίας, όπου έχουμε ένα μεγάλο συνολικό πλαίσιο για σημαντικά προγράμματα και ακόμα περισσότερο από ό,τι για το Connecting Europe είναι ακόμα πιο παρακινδυνευμένο να κάνουμε εκτιμήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Τι θα κάνουμε όμως στην Επιτροπή μας. Υπάρχει το Connecting Europe. Θέλει η Κομισιόν εδώ 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το πρόγραμμα αυτό ή όχι, δεν ξέρουμε. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι <clears throat> οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Μεταφορών έχουν τουλάχιστον τα 47 εκατομμύρια στο μυαλό τους όταν συζητούν για την αρχή του πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Βέβαια αυτό δεν φτάνει γιατί δεν τα έχουμε τα 40 εκατομμύρια. Και αυτό ισχύει και για πολύ μικρότερα κονδύλια και πολύ μικρότερα προγράμματα. Ξέρουμε ότι τα μεμονωμένα προγράμματα τα οποία θέλει να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιβάλλον, όπως το πρόγραμμα LIFE, θα είναι το 1 δέκατο σε χρηματοδότηση από αυτό το οποίο απαιτεί το Connected Europe. Αλλά και εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε για τις βασικές αρχές και ιεραρχίες μεταξύ μας. Και τότε αν πάρουμε τα 3 δισεκατομμύρια ή τα 7 δισεκατομμύρια θα πρέπει αυτά τα κονδύλια να κατανεμηθούν βάσει των αρχών που θα έχουμε θεσπίσει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα αριθμητικά ποσά. Αυτό το καταλαβαίνετε. Ωραία, σίγουρα. Και μετά υπάρχει αυτό που είπε ο Ιβάλλο Καμφίν. Αν εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμών δώσουμε μια γνωμοδότηση σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου δώσουμε τη θέση μας, θα πρέπει να ζητήσουμε και από τις επιμέρους επιτροπές να ζητήσουμε να κάνουν τη γνωμοδότηση για τη δική μας έκθεση. Και τότε είναι φανερό ότι θα πρέπει να έχουν στοιχεία. Αλλά η προκαταρκτική βασική εργασία που κάνουμε τώρα δεν χρειάζεται αριθμός. Giovanni. Καταλαβαίνω πολύ καλά, λέει ο Ρικέ. Αυτό το οποίο λέω, σε ορισμένε περιπτώσει, είπα για το Connecting Europe Facility, για κάποιες περιπτώσεις αλλάζει το περιεχόμενο της ε, απόφασής μας σαν συνάρτηση των κονδυλίων. Αν χάσουμε λοιπόν τα 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής, από το Ταμείο Συνοχή, τότε αλλάζει τελείω η πρότασή μα. Καταλαβαίνω αυτό που λέει η, πρόταση, η πρόεδρο μα. Θα ήταν όμω σόφρο να ζητήσουμε από τι επιτροπέ να επεξεργαστούν, αλλά να ψηφίσουν μόνο όταν έρθουν τα αριθμητικά στοιχεία, ακόμα και αν αυτό είναι καθυστερημένο. Εγώ αλλάζω ιδιότητα και από μέλος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού γίνομαι λίγο το μέλος ε, της Επιτροπής ε, Γεωργίας και αυτού του Financing Cup. με ποιο τρόπο οι εισηγητές προσπαθήσαμε να βάλουμε στην, στην έκθεση ένα recital, ένα εκτιμώντας που λέει ότι τα όσα αναφέρουμε μετά σχετίζονται με το την πρόταση που θα υποβάλει η Κομισιόν για το νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πρόγραμμα. Αν υπάρξουν σημαντικές ε, διαφορές ε, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, είναι προφανές ότι τα όσα έχουμε αναφέρει σε εκείνο το σημείο θα τα ξαναεξετάσουμε. Και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε όλη τη διαδικασία με την παρουσίαση, την υποβολή τροπολογιών, την αναζήτηση των συμβιβαστικών ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες, χωρίς όμως να κάνουμε στην τελική ψηφοφορία για τα νούμερα. Θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία όταν θα δούμε την αντιστοιχία μεταξύ των όσων υπήρχαν μέσα στην πρόταση της Κομισιόν ε, για το Πουδουπού και τα όσα θα είναι τελικά στην, ε, στην τελική συμφωνία. Και θα ξανα, διαφορετικά θα επανέλθουμε και θα ξανανοίξουμε το ντοσιέ και τότε θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ε, Thank Σας ευχαριστώ. Μία επιπλέον ε, πληροφορία. Αποφασίσαμε και θα προτείνουμε στις επιτροπές τροπολογίες που θα είναι οριζόντιες. Δηλαδή, θα ζητήσουμε από όλες τις επιτροπές να υιοθετήσουν τις ίδιες τροπολογίες και η πρώτη λέει ότι ακόμα κι αν μιλάμε για το ε, δημοσιονομικό κονδύλι, δεν θα ψηφιστεί, δεν θα εγκριθεί πριν την υιοθέτηση του, πολιετέ, πλαισίου. Φυσικά και στο πλαίσιο της κάθε επιτροπής θα συζητήσετε τα νούμερα, αλλά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πριν πάμε στην Ολομέλεια να επανέλθουμε στα κείμενο και να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές αφού θα έχουμε πια την εικόνα και τη γενική προοπτική. Θα έλεγα λοιπόν πως ίσως η τελική ψηφοφορία στην Κομισιόν θα πρέπει να γίνει πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάπως αργότερα, δεν είναι ανάγκη να γίνει αμέσως τώρα, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για την νομοθετική βάση με το Συμβούλιο για όλα τα, και για όλα τα άλλα πράγματα και για όλους τους μηχανισμούς. Νομίζω ότι με τη συζήτηση έχει διαλευκανθεί κάπως η κατάσταση. Προφανώς πρέπει να μιλήσουμε πολύ με τις ε, επιμέρους επιτροπές για να καταλάβουν την κατάσταση. Ο κάθε εισηγητής ο οποίος συμμετέχει στην επεξεργασία των νέων δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να τους ε, ζητήσω να είναι παρόν την Πέμπτη το πρωί στο Στρασβούργο που θα κάνουμε μια συνάντηση όλων των εισηγητών και εκεί θα συζητήσουμε όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουν ε, ανακύψει στον τελευταίο μήνα και όλες τις καινούριες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, μήπως θα μπορούσαμε να πάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, αλλά σας παρακαλώ να να το έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε ακόμα την εισηγήτρια για το σημείο 7. Ελπίζουμε ότι στις 4.30 θα είναι εδώ. Και ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε με τον Γιάνν Κοσλόφσκι τότε. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το, ο μηχανισμός αυτός εταιρική ε, σχέσης για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες θα, θα αντικαταστατήσει το 2014 το, ισχύον, τον ισχύοντα μηχανισμό για, ε, για συνεργασία με εκβιομηχανισμένες χώρες και με χώρες ε, με υψηλά εισοδήματα. Η θέσπιση ενός ε, νέου μηχανισμού εταιρικής σχέσης και η χρηματοδότησή του είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι συγκεκριμένη η περίοδος εφαρμογής. Έχουμε στο μεταξύ αναδυόμενες οικονομίες, αλλαγή της δομής του εμπορίου, τη σύναψη νέων και περίπλοκων συμβάσεων και με άλλους εταίρους, όλο και περισσότερες χώρες που αναδύονται και αναπτύσσονται Γι' αυτό και ο νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός μπορεί με αποτελεσματικό τρόπο να προασπίσει τα κοινοτικά συμφέροντα, τα κοινοτικά συμφέροντα στον υπόλοιπο κόσμο. Και το επόμενο ε, επιχείρημα υπέρ του νέου μηχανισμού είναι η ανερχόμενη οικονομική δύναμη χωρών όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία και άρα η ανάγκη ευρυθούς διαλόγου και ε, συνεργασίας με τις χώρες αυτές, κάτι που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής ε, για το 2020. Το νέο αυτό μέσο εταιρική σχέσης ε, θα υλοποιήσει τους εξής στόχους. Θα εξασφαλίσει την ε, διεθνή διάσταση της στρατηγικής του 2020, προωθώντας τον πολιτικό διάλογο και προωθώντας επίσης μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Δεύτερον, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και η διευκόλυση των εμπορικών, ε, επενδυτικών και οικονομικών δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τρίτον, προώθηση της προβολής ε, και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο. Και τέλος, διάλογος και συνεργασία με τις ε, σημαντικότερες από οικονομικές χώρες και τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε και τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Προτείνουμε καταρχήν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα δισεκατομμύριο ευρώ για το 2014-2020 σε σχέση με το ισχύον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ε, κονδύλιο αυτό είναι 304 εκατομμύρια. Βέβαια, για το επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Περιμένουμε τη συμφωνία για να δούμε ποιο ακριβώ θα είναι το ποσό. Θα ήθελα στη δική μου γνωμοδότηση να θίξω τα εξή ζητήματα. Καταρχήν την αναγκαιότητα ενίσχυσης της συνοχής και του συντονισμού ε, στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία εξασφάλιση της χρηματοδότησης, βελτίωση της συνέργειας και της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής χρηματοδότησης. Δεύτερο, στην γνωμοδότησή μου θα ήθελα να τονίσω την ε, ανάγκη υπογράμμισης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψη αποφάσεων αλλά και στην εφαρμογή αυτού του χρηματοδοτικού μηχανισμού. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για δαπάνες ε, του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ε, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ε, συναρμόδια για τον προπολογισμό αρχή είναι σημαντικός. Θα πρέπει να διαλευκαθεί το κατά πόσο θα δημιουργηθεί και ένα αποθεματικό στα πλαίσια αυτού του νέου μηχανισμού. Και αν ναι, ποια θα είναι τα κριτήρια για την ε, κινητοποίηση και χρησιμοποίηση αυτού του αποθεματικού. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ σε ένα σημαντικό σημείο, τον σημαντικό ρόλο που θα έχει στο μηχανισμό εταιρική σχέση η προαγωγή των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η εμφάνιση αυτού του μηχανισμού εταιρικής σχέσης σε καμία περίπτωση θα πρέπει να διαταράξει τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, ούτε θα πρέπει να ε, φέρει σε δυσμενή θέση τις επιχειρήσεις μας ή να παραβλάψει την ανταγωνιστικότητά τους το νέο εργαλείο, αυτό ο νέο μηχανισμό εταιρική σχέσης για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι σημαντικό ε, μέσο για να υλοποιήσουμε τους ε, διεθνείς μας στόχους αλλά και τους στόχους τη στρατηγική του 2020. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ λέει πρόεδρο. Υπάρχουν κάποιες ε, παρατηρήσεις σκιώδεις συζητητέ από άλλε πολιτικέ ομάδε που θα θέλανε να εκφραστούν για το θέμα αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι κάνουμε ανταλλαγή απόψεων εδώ. Για αν φαίνεται ότι τους έχει πείσει όλους. Είναι όλοι σύμφωνοι μαζί σου. Όλα εντάξει, εντάξει, όλα εντάξει. Τα μάμ, τα πάντα εντάξει. Α, ναι, πρέπει να αναφέρω αυτό εδώ τώρα. Εγώ έχω δει την έκθεση μόνο στα αγγλικά, αλλά η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 25 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, όπως πάντα. Ψηφοφορία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 Στις 21 Ιουνίου θα γίνει ψηφοφορία, οπότε εμείς προφανώς πρέπει να δώσουμε τη γνωμοδότησή μας προηγουμένω. Λοιπόν, δεν θέλει κανεί το λόγο, το κατάλαβα και αυτό. Εντάξει. Ja, So, jetzt haben wir ein Problem. Wir sind ohnehin nur noch ganz wenige Abgeordnete hier. Δεν είμαστε πάρα πολλοί ως βουλευτές εδώ ή η η τριά μας. Για το σημείο 7 δεν είναι παρούσα και δεν τη βλέπω να μπαίνει από την πόρα. Μα εδώ είναι, εδώ είναι. Όχι. Μπορείς να μας πεις κάτι για την... Εδώ είναι. Μπορείς να μας πεις κάτι για τα θέματα του δημοσιονομικού κανονισμού στο φάκελο στο φάκελό μου φαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα έρθουν στις 5. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Γέγκλ. Δεν θέλω τώρα να χρειάζεται να τα πούμε δύο φορές επειδή προχώρησαμε πολύ γρήγορα. Αλλά δεν θέλω τώρα και να κάνουμε ομιλίες 10 λεπτών για να καθυστερήσουμε. Ja, das ist, wer weiß, wo die abgeblieben ist. Also, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen gegenüber den... Echo Tipsis Sinidiseon. για του συναδέλφου που του πίεσαν να τελειώσουν. Και επίση και το γεγονό πρέπει να κάνουμε μια διακοπή ενώ είναι πέμπτη απόγευμα. Ναι, Ελίζαμπετ. Ο Γιάν Μίλτερ είναι εδώ παρόν και μπορεί να πει κάτι αυτός από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Είναι ένας εξέχων εκπρόσωπος. Εγώ πάντως είμαι έτοιμη να τα ξαναπώ όταν έρθουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, άμα χρειαστεί. Αν συμφωνούν και όλοι οι άλλοι, ας το κάνουμε έτσι, ας περάσουμε στο σημείο υπαριθμών Τη σημερινή διάταξη και δεν κάνουμε διακοπέ. Έχει το λόγο. Μετά από την τελευταία ανταλλαγή απόψεων εδώ, κάναμε τρει ακόμα τριγωνικού διαλόγου και ο Γιάνν Μίλτον ήταν πάντα παρόν σε αυτέ τι συναντήσει. Έχουμε εξετάσει όλα τα άρθρα, εκτός από το άρθρο 197 και τα άρθρα 206-208 που είναι μεταβατικές διατάξεις και πρόκειται για τις κατεχώρηση κατεξουσιοδότηση πράξη. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα, αλλά οι γενικέ γραμμές, οι αδρές γραμμές, η ακύρωση και η μεταφορά των πιστώσεων, παραμένουν αυτά ανοιχτά, τα προσωρινά 12 τιμόρια και εκεί προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. έχουμε ε, την ε, εναλλακτική λύση που έχουμε καταθέσει με τροπολογίες να μην υπάρχει καθόλου προϋπολογισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψάχνουμε μια λύση για τις μεταφορές, άρθρα 22 με 25, επίσης το άρθρο 29 για τον κίνδυνο σφάλματος και υπάρχουν κάποια άλλα σφάλματα, το 47 ε, και 48, τα μεγάλα κονδύλια, επίσης, η επιμερισμένη διαχείριση και το άρθρο για τις διορθώσεις το 76 και το 77 συγκεκριμένα. Επιμένουμε να υπάρξει σαφής καθορισμός και οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, ενώ το Συμβούλιο θέλει να περιοριστεί σε να περιγράψει τις λειτουργίες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις διορθώσεις στον προϋπολογισμό, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασάφειες. Δεν θέλουμε εμείς λοιπόν να δεχτούμε να γίνει κάτι τέτοιο λόγω της αρνητικής εμπειρίας που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θέλουμε να έχουμε πιο αυστηρές προϋποθέσεις για επιστροφές και εξαιρέσεις. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε την φυσιολογική λειτουργία του προϋπολογισμού. Επίσης το θέμα της πιστοποίησης είναι κάτι για το οποίο διαφωνούμε με το Συμβουλίο. Προβλέπει η Κομισιόν ότι τα κράτη-μέλη πιστοποιούν τις ελεκτικές αρχές, ενώ το Συμβούλιο λέει ότι τις διορίζουν. Ότι τις διορίζει και μετά κάνουν ό,τι θέλουν οι εποπτικές αρχές κατά το Συμβούλιο. Και επίσης στις ε, πληρωμές το Συμβούλιο πιο περιοριστικές προϋποθέσεις για την ε, διακοπή των πληρωμών αλλά πιο αυτόματο τρόπο για να λήγουν οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται. Και επίσης για, το, για τη δήλωση αξιοπιστίας έχουμε μία διαφορά. Είμαστε μαζί με την Κομισιόν εναντίον του Συμβουλίου στο θέμα αυτό και για το θέμα της ετήσιας, του ετήσιου ελέγχου. Τι σημαίνει ετήσιος? Ότι δηλαδή τα προγράμματα θα πρέπει να ελέγχονται μια φορά το χρόνο. Θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όμως σε κάθε πρόγραμμα τι, γίνεται κάθε χρόνο. Θέλουμε κάθε χρόνο να μπορούμε να ελέγξουμε κάθε πρόγραμμα και να δούμε τι έχει πληρωθεί και τι δεν έχει πληρωθεί. Έχουμε τα άρθρα 128-129. Θέλουμε οι τιμές να βρίσκονται σε ένα βασικό, να, ε, να έχουν ένα βασικό επίπεδο 2 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ε, αποδείξεις να δίδονται, ενώ η Κομισιόν λέει 5 εκατομμύρια. Μέχρι 5 εκατομμύρια να μην χρειάζονται αποδείξεις για όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν συνέχεια και έχουν να κάνουν και με θέματα που μας ενδιαφέρουν. Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε κάνει μια σημαντική επεξεργασία και προς το παρόν Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, σε μια θετική συμφωνία. Έχουμε συνδέσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο βασικό δίκαιο. Έχουμε αναφερθεί στα project bonds ως χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Συμβούλιο έχει κρατήσει μια επιφύλαξη στο σημείο αυτό. Επίσης, τα έσοδα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να είναι έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί το Συμβούλιο είναι εναντίον. Εμεί δεν θέλουμε να έχουμε αυτό το εργαλείο μονάχα μια φορά, αλλά από τη στιγμή που δουλεύει. Μήπως μπορείτε να, συ, να εκεί πέρα. Συγγνώμη. Και για την υποχρέωση παροχής εκθέσεων, έχουμε μια καλύτερη εποπτεία που θα έχουμε γιατί θα υπάρχει ένα σχέδιο, ένα έγγραφο το οποίο θα αναφέρει για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία πώς έχουν λειτουργήσει, τι πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα έχουν και τι απόδοση. Αυτό το πρόσθετο έγγραφο εκτός του προπολογισμού θα μας δώσει μια καλύτερη επισκόπηση πέραν των μέχρι στιγμής υποχρεώσεων παροχής εκθέσεων. Επίσης πρέπει να κλείσουμε και το θέμα της πρόορης περάτωσης ενός προγράμματος. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα συναντηθούμε με το Γενικό Διευθυντή του Προϋπολογισμού της Κομισιόν για να επαλέθουμε στο θέμα αυτό. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι προβλήματα που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε για την απαλλαγή. Δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου, ούτε ρούπι δεν έχουμε προχωρήσει. Ειδικέ συνθήκες για τις ερευνητικές θέσεις ειδικά θέματα για να λύσουμε για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. στο τομέα της έρευνας πάντως έχουμε κάνει μια μεγάλη τομή για τους δικαιούχους για να εξασφαλίσουμε κάποιες σημαντικές απλοποιήσεις. Έχει γίνει δεκτό ότι μπορούν να δίδονται ε, πληρωμές κατά αποκοπή και μια καταποκοπή πληρωμή είναι καταποκοπή και δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς χρόνια για να ξαναυπολογιστεί εκ των υστέρων. Για τα θέματα λοιπόν του, των ερευνητικών κονδυλίων έχουμε προχωρήσει πολύ καλά. Για τα καταπιστεύματα <clears throat> θέλει να τα περιορίσει το Συμβούλιο. Εμεί όχι, θέλουμε να δώσουμε στην Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να διαχείριζεται καταπιστεύματα όταν αυτό το θεωρεί απαραίτητο. Θα έχουμε ένα τριγωνικό διάλογο με την ε, Μόνικα επίσης για τα κτίρια και υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα όπου θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Οι εταιρικέ σχέσει δημοσίου ιδιωτικού τομέα έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε κάποια κάποιες που λένε θέλουμε να έχουμε το ευρωπαϊκό υπόδειγμα για τι εταιρικέ αυτές σχέσεις, αλλά όχι να ακολουθούνται τα εθνικά μοντέλα για το πώ θα γίνονται αυτέ οι εταιρικέ συμπράξει Και στο πρόγραμμα πλαίσιο τι θα κάνουμε αν το 1 τρίτο των κονδυλίων τελικά συνδέονται με σχέδια που βασίζονται σε συμπράξεις ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Τότε θα πρέπει να προσδιορίσουμε ήδη το 1 τρίτο των κονδυλίων που δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να ξεδιαλύνουμε το θέμα αυτό των ε, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού. θα πρέπει να ξέρουμε ότι ένα κομμάτι από τον προπολογισμό τότε δεν θα μπορούμε να το επηρεάσουμε. Είναι ένας αυτοματισμός ο οποίος <clears throat> θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σε ετήσιο επίπεδο να επηρεάσουμε και τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ώστε να μην έχουμε ένα μαύρο κουτί μέσα στον προϋπολογισμό για τα ερευνητικά ταμεία. και επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συνδέονται οι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με χρηματοδοτικά εργαλεία και δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση που το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία δυνατότητα να επέμβει στα θέματα αυτά ως αρχή του προϋπολογισμού. Επομένως, εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ικανότητά μας ως αρχή του προϋπολογισμού να επηρεάζουμε πάντα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό με το Συμβούλιο. Η κατεξουσιοδότηση νομικές πράξεις, αυτή τη συζήτηση δεν την έχουμε κάνει ακόμα. Δεν έχουμε προχωρήσει σε περιεχόμενο λεπτομεριακά. Είναι πολλά πράγματα λοιπόν που σας είπα για τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Ποια μορφή έχει το σχέδιο του προπολογισμού, τι έγγραφα συνοδευτικά παραστατικά πρέπει να ε, περιλαμβάνει. Έχουμε κάνει πιο σαφές το πλαίσιο και το έχουμε απλοποιήσει. Και έχουμε καταφέρει να ξέρουμε ποιε είναι οι δέσμε εγγράφων που συνάπτονται σε κάθε, με κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ και έχουμε συμφωνήσει για όλα σχεδόν τα θέματα μέχρι το άρθρο 55. παραμενουν δύο-τρία πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά. το θέμα της διαχείρισης της επιμερισμένης το 56 μένει ακόμα ανοιχτό. Το 57 και το 58 η, ο έλεγχος εξάντε, το 59 η εκτελεστική φορής. Το θέμα του περιορισμού των εξουσιοδιοτήσεων για εκτέλεση του προϋπολογισμού παραμένει αυτό ανοιχτό. Όλα αυτά τα έχουμε μετά το σημείο 72 τους ε, χρηματοοικονομικούς φορείς. Έχουμε λύσει το θέμα της λογιστικής, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την, ε, το λογιστικό έλεγχο, τις ε, προμήθειες. Οι ειδικέ προβλέψεις για την γεωργία, την εξωτερική πολιτική, το πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης, όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διοικητικές πιστώσεις, όλα αυτά τα έχουμε επιλύσει, παραμένουν απλώς μερικές νησίδες αβεβαιότητος και ασάφειας και όποιος θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα εργασίας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αν θέλετε, να έχουμε κάποιους ανθρώπους να έχουμε το πρωί από τις, αύριο από τις 9 στις 3.30 τον ε, τριγωνικό διάλογο και θα πρέπει να δούμε ποια από αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να τα κλείσουμε. Ελπίζω πράγματι ότι στη δεύτερη ολομέλεια του Στρασβούργου θα έχουμε μία λύση και θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε στην ολομέλεια. την ε, Δευτέρα πάλι ξεκινάει ο τριγωνικό διάλογο. Δεν ξέρω αν θα έχει τελειώσει όμω εγκαίρω για να προλάβω να πάω σπίτι μου το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι εκτιμούν το πόση εργασία έχεις κάνει. Λοιπόν, σίγουρα ξέρω πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρεις ότι εγώ σίγουρα δεν θα μπορούσα να κάνω τη δική σου εργασία. Ούτε θα ήθελα να την κάνω. Ούτε θα μπορούσα να την κάνω τη δικιά σου εργασία. Να θέσω όμως ένα ερώτημα μονάχα. Όταν λες ότι κάτι έχει ήδη ότι έχει κλείσει, λες ότι εκεί το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν έχουν αποφασίσει ποια μορφή θα έχει μια συγκεκριμένη παράγραφο στο δημοσιονομικό κανονισμό. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό. Κανείς δεν έχει πει όχι σε κάποιο σημείο. Δεν σημαίνει ότι έχουν πει όλοι ναι. Έχω πάλι ένα ερώτημα. Γιατί αυτό θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τα διάφορα ταμεία. Υπάρχει στο δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος τώρα αναδιαμορφώνεται. Υπάρχουν κάποιες πρόνοιες για την επιστροφή του ΦΠΑ. Ωραία. Μπορείς να μου πεις πώς δουλεύει αυτό. Είναι μία ακόμα από τις παραγράφους που παραμένουν ανοιχτές. Έχουμε θεσπίσει σαφείς κανόνες όπου λέμε ότι ο ΦΠΑ να μην επιστρέφεται. Δηλαδή, όταν ένα κράτος εισπράττει ΦΠΑ, ε, τότε αυτός θα πρέπει να δίδεται στην Κομισιόν και η Κομισιόν έχει προτείνει μια λύση η οποία είναι πάρα πολύ ευφυής. Το Συμβούλιο έχει κρατήσει στάση επιφύλαξη αλλά νομίζω ότι μπορεί να περάσει αυτό το σημείο και εγώ έχω κάποια αισιοδοξία. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Παραμένει ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο που τον αγνοούμε, το θέμα της, του, του ΕΤΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, παραμένει ανοιχτό. γι' αυτό τον ελέφαντα τώρα δεν μπορώ να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποιο, κάποια εξέταση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όμως τον ελέφαντα εκεί πέρα να αλωνίζει. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση για αυτό που αναφέρεις για το ΦΠΑ, δεν μπορούμε να αφήσουμε να χάνεται ο ΦΠΑ στα κονδύλια της, Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Σαλβαδόρ και η Άιντα. Eh, Ευχαριστώ. Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στην Ίγκε και το έργο που επιτελεί. Έχω μία ερώτηση. Όλο και περισσότερο στο, Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούμε για την πιθανή αλληλεγγύη, ε, συγγνώμη, ό,τι αφορά τι μεταφορέ στα τέλη του έτους. Όπως ξέρει, Σίγκε, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τους λογαριασμού του τελευταία στιγμή. Η Επιτροπή λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει τις μεταφορές μεταξύ 31 Δεκεμβρίου και το πρώτο τριμήνο του επόμενου έτους για να πληρώσει αυτούς τους απλήρωτους λογαριασμούς. Γι' αυτό και σκεφτόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει περισσότερη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού, προκειμένου να γίνονται οι διάφορες μεταφορές από χρόνο σε χρόνο. Δεν ξέρω, Ίγκε, το θέμα αυτό της ελαστικότητας αποτελεί θέμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΑΕΝΤΑ. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις προς την εισηγήτρια. Ποιες θα είναι οι επόμενες συναντήσεις, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα του τριμερούς πολιτικού διαλόγου, ποια θα είναι η διάρκεια αυτού του διαλόγου και ποια θα είναι τα θέματα στους μελλοντικούς αυτούς τριμερείς πολιτικούς διαλόγους ποιες είναι οι προθέσεις της συγκεκριτήριας, ποια είναι τα θέματα που εκείνη θα τονίσει ως πιο σημαντικά, ποια ζητήματα είναι πιο προβληματικά. Θέλω κάποιες πληροφορίες για το μέλλον αυτών των τριμερών πολιτικών διαλόγων. Πρωτού κλείσω λοιπόν, δίνοντας το λόγο στην Ίγκε, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν θέλουν να κάνουν μια δήλωση για τις ε, διαπραγματεύσεις σε σχέση με το δημοσιονομικό κανονισμό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η κυρία Γκρέσλε παρουσίασε την κατάσταση πολύ αντικειμενικά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, χάρη στην εργασία της κυρίας Γκρέσλο και των συναδέλφων της Προεδρίας, έχουμε κάνει πρόοδο σημαντική και κυρίως ανοίξανε κάποιες οδοί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όπως είπε, το πιο λεπτό ζήτημα είναι όντως το θέμα της ε, κοινή διαχείρισης. Η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να ευνοήσει την εξέβρεση συμφωνίας ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και νομίζω πως έτσι ανοίξαμε κάποιες προοπτικές. Ελπίζω ότι θα είναι αποδεκτές. Μένει επίσης το θέμα των ε, reflows για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Και τώρα το θέμα του ΦΠΑ πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστεί μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού και επανέρχεται μάλιστα στις συζητήσεις για τους θεμεακού ε, κανονισμούς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά πιστεύουμε πως το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού και με χαρά άκουσα που είπε η κυρία Γκρέσλο ήταν ευφυής η πρόταση της Κομισιόν. Είναι πραγματικό ε, κομπλιμέντο αυτό. Ε, το θέμα της εταιρική σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ναι, ναι, είμαστε συνηθισμένοι. Όχι, είμαστε συνηθισμένοι, αλλά κάποιες φορές ακούμε και αντίθετες, αντίθετα σχόλια. Συνήθως ξεχνάμε τα καλά λόγια και μας μένουν στο μυαλό οι επικρίσεις, γιατί θέλουμε πάντοτε να κάνουμε ακόμη, να τα πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα. Υπάρχει το θέμα των εμβασμάτων. Για τα εμβάσματα υπάρχει μια πρόταση της Κομισιόν και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι το ανέφερε τι προάλλες. Όπως και πέρυσι, ε, βρισκόμαστε σε μια πολύ παράξενη κατάσταση ότι πρέπει να επιστρέψουμε 375 εκατομμύρια ευρώ στα κράτη-μέλη, ενώ αν είχαμε, καν, μια διαδικασία που να μας επέτρεπε να μεταφέρουμε αυτά τα χρήματα, θα είχαμε στο τέλος του έτους 375 εκατομμύρια επιπλέον ως πιστός πληρωμών που θα μας, έπρεπε, θα μας επέτρεπε να χρηματοδοτήσουμε τα ράλα. Δεν είναι τα 5 δις που χρειαζόμασταν, αλλά θα ήταν τουλάχιστον 375 εκατομμύρια. Αυτά είναι ακόμα υποσυζήτηση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια μέθοδο που θα σεβαστεί τα δικαιώματα των δύο σκελών της Δημοσιονομικής Αρχής. Εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κονδύλια που είναι στη διάθεσή μας με σεβασμό στην δημοσιονομική διαδικασία αλλά γνωρίζοντας επίσης πως υπάρχουν προθεσμίες που είναι περιοριστικές. Αλλά πιστεύω πως έχουμε ενδιαφέρουσες προοπτικές αν βασιστούμε και πιο συγκεκριμένα στα προηγούμενα που έχουμε στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχει τέλος και το θέμα που το τελευταίο που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για το πνεύμα το ομαδικό με το οποίο εργάζεται. Συνεργάζεται με την Κομισιόν και νομίζω πως χάρη σε αυτή την πολύ πολύ όμορφη συνεργασία θα μπορέσουμε να έχουμε πια γρήγορα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε πως η Δανική Προεδρία σε πολιτικό επίπεδο θα είναι διαθέσιμη ώστε να γίνουν οι τριμερείς διάλογες σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει όντως να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις πριν το καλοκαίρι, γιατί μετά έχουμε εσωτερικά μια ολόκληρη περίοδο μεταγραφής όλων αυτών των αλλαγών του δημοσιονομικού κανονισμού στα εργαλεία διαχείρισης, δηλαδή στη πληροφορικά μέσα και δεν γίνεται αυτά εν μία νυχτή. Είναι μια πολύ, ένα πολύ βαρύ έργο και άπαξ και δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι συμφωνίες, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά όσον αφορά την προσαρμογή των εργαλείων διαχείρισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ τώρα, αν μπορώ να σας συγχαρώ, για την αγαστή συνεργασία εισηγήτρια και κομισιόν ή αν θα πρέπει να ανησυχήσω. Η Ίγκε, για να κλείσει τη συζήτηση. Μην ανησυχείς. Δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου αυτή. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα και την ομάδα του, γιατί είναι πράγματι πολύ σημαντικά να υπάρχει, να υπάρχει τακτική επεξεργασία των θεμάτων αυτών αυτό το τεράστιο θέμα με πάνω από 300 τροπολογίες δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε χωρίς, μια, τη βοήθεια της επαγγελματικότητας της ομάδας της ε, Κομισιόν και ελπίζω θα μπορέσουμε να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν θέλω να περιμένουμε την επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου και να πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή την επεξεργασία του θέματος αυτό Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την, ε, τον Γιένς για τις προσπάθειές του. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε διαφορές για τα θέματα αυτά. Τώρα τι θα γίνει με τις μεταφορές στο τέλος του χρόνου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και εγώ το αναγνωρίζω και πάλι δίνω ένα δεύτερο κομπλιμέντο στο Γενικό Διευθυντή της Κομισιόν. το... Είχε βρει και εδώ μια ευφυή λύση θα εφεύρουμε ένα 13ο μήνα για να καλύψουμε αυτές τις ε, μεταφορές. Αυτό έχει γίνει ήδη στην ε, Γεωργία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επαρκή ευκαμψία στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή, παρατείνουμε ουσιαστικά τον τελευταίο μήνα. Βρίσκουμε λοιπόν τη δυνατότητα να έχουμε ένα πρόσθετο μήνα μέσα στον οποίο μπορούν να γίνονται αυτές οι μεταφορές. Το Συμβούλιο έχει βέβαια τις αντιρρήσεις του, αλλά εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν. Θα είναι χειρότερα τα αποτελέσματα εάν δεν έχουμε αυτό το τέχνασμα. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά για το τέλος του χρόνου. Είναι ακριβώς ένα σημείο από τα οποία το Συμβούλιο δεν συμφωνεί μαζί μας και χρειαζόμαστε μια πολιτική τομή από την πλευρά του Συμβουλίου για να έχουμε την υποστήριξή του, για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Αυτό σίγουρα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τον πολιτικό τριάλογο, τριγωνικό διάλογο, ή τα ποσά τα οποία ε, μεταφέρονται και πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα με ένα 13ο μήνα, πιστεύω εγώ. Επίσης, το θέμα του ΦΠΑ θα πρέπει να επιληθεί. Εγώ φυσικά θα ήθελα να λύσουμε όσο το λιγότερα προβλήματα με πολιτικό τρόπο, γι' αυτό προσπαθώ να εξεύρω τεξ, τεχνικές λύσεις. Είναι μια λεπτομεριακή εργασία, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι λεπτομέρειες. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα μπορέσουν οι διπλωμάτες της Κορεπέ να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα λεπτομεριακά θέματα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ενδιαφερθούν και μπορούμε να κινδυνέψουμε να έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα σε όλα αυτά. Πρέπει όμως να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που θα εξετάσουν λεπτομεριακά όλα αυτά τα θέματα προηγουμένως ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Γιατί φοβάμαι την, τον τριγωνικό διάλογο αν δεν υπάρχει πραγματική θέληση από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρξει κακό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλω κάθε φορά να πηγαίνουμε με ένα μικρό αριθμό θεμάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ μακρύ κατάλογο θεμάτων τα οποία υπόκεινται στον ε, τριγωνικό διάλογο και θα πρέπει κάθε φορά να παρουσιάζουμε μονάχα μερικά από αυτά τα σημεία ώστε να μπορούν και οι εκπρόσωποι της Κορεπέρ να εγκρίνουν αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι η θέληση να προχωρήσουμε υπάρχει οπωσδήποτε από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά του Κομισιόν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πάντως τον πολιτικό τριγωνικό διάλογο, να κάνουμε τις προσπάθειες για να βρούμε λύσεις. Δεν είναι θέματα ουσίας μονάχα, είναι και θέματα πολλές φορές αποχρώσεων και προσέγγισης είναι μια πρόκληση να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και έχουμε στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό νέα στοιχεία. Χρηματοδοτικά εργαλεία, καταπιστεύματα, σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα είναι καινούργια σημεία για τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια, ένα αριθμιστικό πλαίσιο, ένα κανονιστικό πλαίσιο και πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους κανόνες και τώρα αν αυτοί οι κανόνες <clears throat> αποδειχθούν ότι δεν είναι πρόσφοροι θα πρέπει σε δύο χρόνια να επανέλθουμε. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε την Ίγκια για την πολυσχηδή της εργασία. Και ερχόμαστε τώρα και σας λέμε μέχρι την επόμενη έκθεσή σας. Το τελευταίο σημείο της ημέρας διάταξης, το λουκούμιο σημείο, των υπαριθμών 7 κ. Γιένσκι είναι παρόν πλέον και μπορούμε να σταθούμε στην ετήσια έκθεση του Συμβουλίου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ και κυρίως ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Το εκτιμώ όλος ιδιαίτερος. Θα περάσω αμέσω στην ουσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην γνωμοδότηση του προπολογισμού για την ετήσια έκθεση ΚΕΠΑ για το 2010 καλωσόρισα τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της ευρείας συλλογής μέσων που χρησιμοποιεί και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της περαιτέρω βελτίωσης του συντονισμού ανάμεσα στα διάφορα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στρατηγική, πολιτική πολιτικά σκέλη ε, δεδομένων των περιορισμένων πόρων που έχουμε στη διαθεσή μας για την ΚΕΠΑ και άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, όλες οι δυνατότητες και να υπάρξει ο μέγιστος συντονισμός. Σε αυτή την ε, περίοδο η ΚΕΠΑ είναι υπό έναν ex post έλεγχο, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των νέων προτάσεων για τους νέους κανονισμούς για την εξωτερική δράση. Καταρχήν αναγνωρίζω το γεγονός ότι παρά τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της ΚΕΠΑ, το αποτέλεσμα το 2010 ήταν μόνο 282 εκατομμύρια ευρώ, είτε 3,5% της συνολικής ε, των συνολικών κονδυλίων για την κατηγορία 4. Θα σας θυμίσω επίσης το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο στρατηγικά περιόρισε τα κονδύλια για την ΚΕΠΑ εγκαίρως πριν από την ε, ε, συνεδρία της συνδιαλλαγής πέρσι. Θα αφήσω τη στρατηγική τη φετινή για τις περαιτέρω συζητήσεις, αλλά θα ήθελα να έχετε υπόψη σας όλα αυτά όταν συζητάμε ε, για πιθανές ε, συνεργασίες. Ε, μπορεί να έχουμε λόγο να περιορίσουμε τον, περιορισμό, τον προϋπολογισμό αν δούμε κάποιες διαφορές ανάμεσα στα ποσοστά απορρόφησης για την υπερσινή χρονιά σε αντίθεση με την κατανομή των υποχρεώσεων για το 2012. Ο κύριος Λαμασούρα έχει στείλει επιστολή για να ρωτήσει γιατί οι γραμμές της ΚΕΠΑ που δεν απορροφήθηκαν το 2011 αυξήθηκαν περισσότερο στα κονδυλιά τους για το 2012. 12 με 3 με 5 φορές μεγαλύτερη αύξηση από ότι κάποιες γραμμές οι οποίες εξήλυσαν τις πληρωμές τους. Ελπίζω πως θα λάβουμε κάποιες απαντήσεις για αυτό το ενδιαφέρον θέμα που αφορά τον ε, προγραμματισμό και συγχαίρω τον κύριο Λαμασούρ παρότι λείπει αυτή τη στιγμή για την ε, δραστήρια εμπλοκή του. Να σας πω τώρα τι έγινε στις συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με τη μελέτη της κόστους αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Τα ποσά τα οποία δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για την πρόληψη συγκρούσεων και για τη διαχείριση κρίσεων θα έπρεπε να μετακινηθούν περισσότερο προς το ε, επιχειρησιακό ε, οδηγό γιατί λείπει ναι, ο συντονισμό ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και οριζόντια ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια, πράγμα που είναι απαραίτητη προπόθεση ώστε να υπάρξουν ε, συνέργειε ε, από κάτω προ τα πάνω, όπω για παράδειγμα στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη. Πού μπορούν να γίνουν βελτιάσει. Καταρχήν, μεγαλύτερη συγκέντρωση και κατανομή των, κυρί... των στρατιωτικών δυνατοτήτων, βελτίωση των δυνατοτήτων για σχεδιασμό επιχειρήσεων, ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών αποστολών και επίσης νομίζω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι παρουσιάσεις για το κόστος και για τη διαφάνεια θα πρέπει να προηγηθούν οποιονδήποτε άλλων βελτιώσεων όσον αφορά τις ευρωπαϊκές δυνατότητες. Γι' αυτό και έχω προτείνει έναν κανονισμό με, όπου θα έχουμε συγκεκριμένη γραμμή για κάθε μία αποστολή ΚΕΠΑ και έτσι να έχουμε μία σαφή εικόνα για τις αποστολές. Ο μηχανισμός για τη χρηματοδότηση του κοινού κόστους των ε, στρατιωτικών και αμυντικών επιχειρήσεων της Ένωσης δεν μας δίνει επαρκή εικόνα για τις ε, οικονομικές επιπτώσεις των ε, αποστολών που γίνονται υπό την ΚΕΠΑ. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κανείς να λάβει το λόγο σχετικά. έχει επέλθει κάποια κόπωση επειδή είναι πέμπτη απόγευμα. Και όλοι αυτοί που έχουν μείνει εδώ πέρα έχουν στα μάτια τους το Πάσχα και τον Οβελία. Σας λέω λοιπόν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 25 ε, Απριλίου το μεσημέρι όπως πάντα και η γνωμοδότηση θα ψηφιστεί στις 31 Μαΐου και θα τη στείλουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που θα ψηφίσει τον Ιούνιο, αν θέλει ο Θεός. Αν δεν θέλει κανείς να κάνει σχόλια για την πλήρη έκθεση της Ναζδέσδα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της συνεδριασής μας. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι άντεξαν ως το τέλος και σας εύχομαι ευτυχισμένο Πάσχα και κάποια ξεκούραση την επόμενη εβδομάδα η οποία είναι χρώματος τυρκουάζ. Θα τα πούμε τον Απρίλιο.